Good morning, colleagues from... Συνάδελφοι, καλημέρα και από τις δύο επιτροπέ. Θα ήθελα μαζί με τον Συμπρόεδρο κ. Λάγκε να σας καλωσορίσω στην κοινή μας συνεδρίαση των δύο επιτροπών για να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης για την ισότητα των φύλων εντός των ε, εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης. Ο λόγος στον Συμπρόεδρο. Καλημέρα και από μένα συνάδελφοι. Είχαμε μια κοινή προσπάθεια μεταξύ των δύο επιτροπών μας, ΦΑΜ και ΙΝΤΕ, και είχαμε ένα πολύ θετικό διάλογο με πνεύμα συνεργασία και από τους δύο. Τελικά έχουμε την έκθεσή μας με πάνω από 300 τροπολογίες και νομίζω 43 συμβαστικέ προτάσεις ώστε να τις ψηφίσουμε σήμερα. Μεγάλη ψηφοφορία έχουμε μπροστά μα σήμερα, έτσι. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα πρέπει να τροποποιήσουμε την ημέρησια διαταξή μας, αν χρειάζεται. Αν δεν υπάρχουν, θεωρείται εγκεκριμένη. Δεύτερο σημείο στην ημέρησια διάταξη είναι η έκριση των πρακτικών του Νοέμβρη του 2017. Δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια παρατηρήσεις, συγκρίνονται τα πρακτικά. Και τώρα θα ξεκινήσουμε την ηλεκτρονική μας ψηφοφορία. Να έχετε τις κάρτες σας έτοιμες, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Ε, gender equality in... Η ισότητα λοιπόν των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, έκθεση Φορέντσα και Μπιόρκ και θα ξεκινήσουμε τώρα την ηλεκτρονική μας ψηφοφορία με τη συμβαστική πράξη 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 20 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 λέει πρόεδρος υπέρ κατά αποχές πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται ναι παρακαλώ δεν έχω την κάρτα μαζί μου. Μπορώ να ψηφίσω δια ανατάσεως. Ναι, βεβαίως. Μαρία, μπορείς. Όχι όμως ίσως την προσωπική ψηφορία. Μπορεί ενδιάμεσα να πας να ζητήσεις την κάρτα σου. Γίνεται, μπορείς. Ωραία. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω εγκρίνεται, αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Περάς. Yes. Yes. Εγκρίνεται. Is in Και η Μαρία είναι υπέρ. Και η Μαρία είναι υπέρ. Yeah, Maria is in favor. Η Μαρία λοιπόν είναι υπέρ. yeah, she has forgotten the voting card, but. Είχε ξεχάσει και την κάρτα της η Μαρία. Θα ξαναρχίσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. 190, 190 ξαναψηφίζουμε. Άρχεται πέρας. Πέρας ξαναλέει πρόεδρος. Yes. Yeah. Okay. It will be done. Ωραία. Τελευταία φορά, έτσι. Τελευταία φορά που θα ξαναψηφίσουμε. Το λέω να το ξέρετε. <laughs> Για την 190. Τελεία και παύλα, συνάδελφοι, έτσι. Τελευταία φορά, ξεκινάμε τώρα, τελευταία φορά ψηφίζουμε, να το ξέρετε. Ψηφίσατε όλοι. Ρωτάει ο πρόεδρος δυνατά. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 191. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 199 ως προσθήκη στη συμβαστική 25 υπέρ. Κατά, άποχες, εγκρίνεται Συμβιβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. 203. 203. Άρχεται. Πέρας τώρα. Απορρίπτεται. 28 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 217 υπέρ. Η πρώτη καταλάβωση είπε 2017. Είναι 2017. Διορθώνει τώρα Συγγνώμη λέει η πρόεδρος, είχα πει 2017. Συγγνώμη λέει. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Και τώρα πέρας. Απορρίπτεται. 2.18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να αλλάξουμε. Εντάξει. Για, το 200, για την 218 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...232 υπέρ... ...υπέρ, ξαναλέει πρόεδρος... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται... 230. Πέντε πήγε να πει πρόεδρος. Όχι, όχι, λάθο λάθο λέει τώρα. Συγγνώμη. Ε, ναι, ναι, επειδή κλπ. κλπ. 233 υπέρ. 233 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. Α, θα ελέξουμε θα έλέξουμε για 234. Άρχεται. Άρχεται για 234. Πέρας. Απορρίπτεται. 235 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέξουμε. Για τη 237 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία και τώρα πέρας λέει πρόεδρος απορρίπτεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 245 υπέρ κατά αποχές θα ελέξουμε για την 245 άρχεται η ψηφοφορία και τώρα πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 246 in favor 246 θα ξαναψηφίσουμε, λέει ο Πρόεδρος. 2.45 για 245. Ξαναψηφίζουμε για 245. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία για 245. Απορρίπτεται. Ε, Συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία μας, έτσι, θα συνεχίσουμε. 246 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 257 ε, σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε, να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται και τώρα πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 261. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ. Κατά. Άποχες. Να ελέξουμε Παρακαλώ άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία και τώρα πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, θα ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε για 272. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, ε, now, amendment 277. 277 υπέρ. Όχι, όχι, καταπίπτει, καταπίπτει λένε της Πρόεδρου. Ε, sorry. Ε, όχι, συγγνώμη, ναι, ναι, καταπίπτει. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ...305 υπέρ... ...κατά αποχές εγκρίνεται... ...309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 182 ως προσθήκη στην συμβαστική 39 υπέρ, κατά αποχές πρέπει να ελέξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 σε τρία τμήματα. 60 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. «318 υπέρ κατά αποχέ. θα ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται πέρας Εγκρίνεται. Ε, Συμβαστική 41 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 331 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. 334 υπέρ. Κατά. αποχέ. πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. It's 42. Απορρίπτεται. 42. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, κατά Κατά πίπτη λέει τώρα ο Πρόεδρος. Amendment 3 in favor. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πέντε και έξι από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές να κάνουμε παλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία πέρας αυτής απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ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 Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. αποχέ, Πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Παρακαλώ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας αυτή, Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτή Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχο καλά λοιπόν. Απαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρχεται η ψηφοφορία για έλεγχο. Πέρας. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Εντάξει λοιπόν, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93. Μόνο αυτό το εδάφιο που περιλαμβάνεται στο ε, δεξί τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, παρακαλώ να επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Απορρίφθηκε. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα 98 μόνο το τμήμα που περιλαμβάνεται πάλι στο δεξί τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρασε αυτή τώρα. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106. Υπέρ, κατά, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Έλεγχο. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρχεται η ψηφοφορία για έλεγχο. 136 ε, πέρας. Με συγχωρείτε, εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Εντάξει, λοιπόν, να σε παληθεύσουμε και την συμβαστική 17, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίθηκε. Υπέρ. Δεύε 15 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύε 17, δεύτερο τμήμα, σωστά. Α, καταπίπτει. Κατέπεσε. Δεύε 18 υπέρ. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Δεύε 17 μόνο εκεί που λέει ε, δίνει έμφαση στην ανάγκη συμπεριλαμβανομένη τη ε, ισότητα των φύλων. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίθηκε. Καλά, σε παληθεύσουμε η ψηφοφορία. Και τώρα πέρασε αυτή. Ντέβε 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε αυτής. Απορρίφθηκε. Ντέβε 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε αυτής. Απορρίφθηκε. Δεύε 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ψηφίσουμε. περασε Εγκρίθηκε. Δεύε 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΔΕΒ 25, άρχεται η ψηφοφορία. Και τώρα τελείωσε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. ΔΕΒ 5. Μόνο αυτό που είναι εντό εισαγωγικών. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕΞΙ υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Απορρίφθηκε. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης, έκθεσης μάλλον ως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Μπορείτε να μην ψηφίσετε. Υπάρχει ένας υπεράριθμος. Πέρας τώρα της ψηφοφορίας. Α, εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε, μπράβο. Thank you very much for both. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ καλά η ψηφοφορία, καλή επιτυχία. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία μα. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ. κύριοι βουλευτές. Θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Η Επιτροπή Γενικών θα συνεχίσει